τις οικογένειες και τους Οικείου ε, των ε, θανών των στρατιωτών που θυσίασαν τη ζωή τους για την συμφιλίωση των κοινοτήτων, ε, για την ευημερία των κοινοτήτων αυτών, καθώς και των άλλων θυμάτων Πρόκειται για την πρώτη επίθεση στη Βόρεια Ιρλανδία ύστερα από 12 έτη, ένα βαθύτατο πλήγμα, βαρύτατο πλήγμα κατά των δημοκρατικών θεσμών και τη δημοκρατική κοινωνία τη Βόρεια Ιρλανδία και των πολιτών τη. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στη Βόρεια Ιρλανδία είδα είδαειδή ισόμαση Ε, το πλούσιο μέρισμα θα έλεγα που προσέφερε η συμφιλίωση στη Βόρεια Ιρλανδία και που επιτρέπει στους πολίτες και των δύο κοινοτήτων να οικοδομήσουν από μαζί ένα καλό μέλλον για τις ζωές τους και για τα παιδιά τους. Οι τρομοκράτες που διέπαιξαν αυτό το έγκλημα προσπαθούν να ανατρέψουν τις ψυχολογικές συνθήκες ζωής στη Βόρεια Ιρλανδία, δεν έχουν καμία υποστήριξη στη λαϊκή βάση και η ευρύτατη πλειονότητα των πολιτών τους καταδικάζει. Εκφράζουμε την ελληνική μας στους πολίτες της Βόρειας Ιρλανδίας και στις δυνάμεις ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη αυτού του εγκληματίες. Εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι καταδικάζουμε σε η ανδήποτε μορφή και αν αυτή εκδηλώνεται την τρομοκρατική βία. Οι φόνοι αυτοί δεν θα επιτύχουν την ε, αποδιάρθρωση της δημοκρατικής ε, και ειρηνευτικής διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία, μια ειρηνευτικής διαδικασία στην οποία ανέκαθεν και στεναρά υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο ηθικά όσο και υλικά έχουν επιλέξει ο λαό της Βόρεια Ιρλανδία το μέλλον τη ειρήνη και της αμοιβαία αναγνώριση και σεβασμού τη ε, ε, αξιοπρέπεια του εταίρου για το μέλλον. Και εμεί υποστηρίζουμε την επιλογή αυτή, την επιλογή τη ειρήνη, τη Δημοκρατία, του Κράτου δικαίου και στεχόμαστε στην πλευρό του λαού της Βόρειας Ιρλανδίας αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σα καλέσω τώρα μαζί μου να τηρήσουμε ένα ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των φωνευθέντων στρατιωτών. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ. Ο ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Σάββατο το βράδυ στη Βόρεια Ιρλανδία όλοι και νομίζω ότι μιλώ για λογαριασμό όλων αισθανθήκαμε ε, αποτροπή με, τον, ε, με την αποτρόπαιη και ψυχρό αυτή δολοφονία. Ε, μιλάμε για τον χειρότερο εφιάλτη ε, στην Βόρεια Ιρλανδία. Ε, είμαι μέλος του Κοινοβουλίου για, σχεδόν 20 χρόνια τώρα και ήλπιζα ότι ποτέ πια δεν θα έπρεπε να, σταθώ σε αυτό το Κοινοβούλιο και να προσφέρω τα ε, συλληπιτήριά μου στις οικογένειες ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη Βόρεια Ιρλανδία. Αισθάνομαι ιδιαίτερη λύπη για το γεγονός ότι είμαι αναγκασμένος να το πράξω σήμερα. Αυτοί οι νεαροί άνδρες έπραξαν ε, αυτό το οποίο κάνουν πάρα πολύ ε, συνηθισμένοι νεαροί ε, ε, ε, πραγματικά δεν τα κατάφεραν να επιζήσουν και οι σκέψεις μας είναι σε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα που, τους, που έχασαν τη ζωή τους στο άνθος της τους. Δεν ήρθε η ώρα να πούμε τίποτα άλλο σήμερα παρά μόνο να προσφέρουμε τη συμπάθειά μας στις οικογένειές τους. Αυτή τη στιγμή οι οικογένειές τους χρειάζονται την υποστήριξη αυτή και Βεβαίως, ε, δεν ε, ε, είτε καταδικάσουμε είτε όχι την πράξη αυτή, οι υπέτειοι δεν πρόκειται να συγκινηθούν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρόκειται να πετύχουν, δεν πρόκειται να κερδίσουν τίποτα, γιατί θα κερδίσει η δημοκρατική διαδικασία στην Ιρλανδία. Ε, αυτή τη στιγμή ε, ο λαός μας στη Βόρεια Ιρλανδία ε, ζει μια καλύτερη ζωή. Έχει την εμπειρία αυτή τη καλύτερη ζωή και θέλω να συνεχίζουν να ζουν αυτή την καλύτερη ζωή. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω και εγώ τα λόγια συμπάθεια και συλληπιτηρίων προ τι οικογένειε των ανθρώπων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δύο ακόμη συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο από πλευράς των Βόρειο Ιρλανδών, Ιρλανδών βουλευτών. Κύριε Σόλγουρτ, παρακαλώ. Άιλουρτ ίσω, παρακαλώ. Πρόεδρε, και εγώ καταδικάζω περίφραστα το φόνο δύο στρατιωτών, τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη πολιτών και στρατιωτών που έλαβε χώρα την, ε, το Σαββατοκύριακο αυτό το, το Σάββατο στην περιοχή του Μπέλφαστ. Βλέπουμε ότι οι τρομοκράτε αναλαμβάνουν και πάλι δράση. Ει βάρο των δυνάμεων ασφαλεία, είχαν περάσει 12 χρόνια για να εμφανιστεί άλλη μια τέτοια τρομοκρατική επίθεση. Πρόκειται για φρικτά εγκλήματα, εγκλήματα τα οποία δεν εξασφαλίζουν την πολιτική υποστήριξη των πολιτών τη Βόρεια Ιρλανδία. Η Συμφωνία του 1988 τη μεγάλη παρασκευή, προσδιορίζει ένα σαφέ πλαίσιο οικονομική και πολιτική ανάπτυξη στη Βόρεια Ιρλανδία και βάσει αυτή τη συμφωνία τη Μεγάλη Παρασκευή εργάζεται ο κόσμο για να αναπτύξει τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου, την ειρήνη και τη συμφιλίωση, την επανασυμφιλίωση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε λοιπόν σε τέτοιου είδου άτομα να πλήξουν την ειρήνη για την οποία τόσο πολύ αγωνιστήκαμε όλοι στη Βόρεια Ορλανδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Ράιν Ερβουλτ και ο Τζι Ellison, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σε ευχαριστώ ε, για τα ε, λόγια σας ε, προς τους ε, των νεαρών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο το βράδυ. Και πράγματι πρέπει να σκεφτόμαστε όλους αυτούς που πενθούν αυτή την κρίσιμη στιγμή. Θα ήθελα να πω ότι οι πέτοι της δολοφονίας αυτών των στρατιωτών θέλουν να, θέλουν πολιτικά ωφέλη μέσω του δρόμου της βίας. Θέλω να πω ότι δεν πρόκειται να πετύχουν το σκοπό τους. Δυστυχώς όμως στη Βόρεια Ιρλανδία φαίνεται ότι τελικά ε, η βία είναι ένα ε, φαινόμενο που, ε, που ανταποδίδει, διότι σήμερα τρεις πρώην καταδικαστέντες συμμετέχουν στην κυβέρνηση και ε, ε, και μάλιστα για, ε, για ορισμένους, ορισμένους είχε αναφερθεί η κατηγορία ότι είχαν σκοτώσει 12 ανθρώπους. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καλύτεροι από τους υπόλοιπους τρομοκράτες οι άνθρωποι αυτοί. και μάλιστα ε, ε, κάποιος ο οποίος είχε, ε, είχε περιγραφεί ως ε, χασάπης, ως αποτρόπος δολοφόνος. Και όμως ε, αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν όταν διαπραγματεύεται κανείς με τους τρομοκράτες. ελπίζω όμως να μην ξανασυμβεί στο, στο μέλλον και να διδαχθούμε τα διδάγματα του παρελθόντος και να μην φερθούμε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ. Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι Αυτά. Δεν μπορούμε τώρα κάθε Ιρλανδό βουλευτή να παρακαλέσουμε να παρέμβει. Να παρέμβει αναφέρθηκαν αυτές οι παρεμβάσεις εξ ονόματος και των άλλων. Συμφωνείτε ότι με αυτόν τον τρόπο είχαμε μια σωστή απότηση φόρου τιμής ε, στους δολοφονημένους στρατιώτες. Εντάξει. Και μια σύντομη δήλωση για την ημέρα των γυναικών εχθές. Με αυτή την αφορμή θα ήθελα όλους τους ε, συναδέλφους ε, να τους χαιρετήσω στην, Ευρω... στην Ευρωβουλή και να ευχαριστήσω ρητά και κατηγορηματικά για την προσπάθεια που έγινε και θέλω να πω ότι Κάθε προσπάθεια γίνεται ώστε η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των φύλων ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια να μπορέσει να υλοποιηθεί. Πριν από 100 χρόνια